και τώρα περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου, συνάδελφοι. Αρχίζουμε με τον προϋπολογισμό του 2012. Ο κύριος Φόξ θέλει να μας εξηγήσει πώς εψήφισε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η σημερινή ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό είναι άλλη μια χαμένη